ΠΠΕ, ΕΛΚ, ECR, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες και e ΕΝΕΦ και οι μη εγγεγραμμένοι βουλευτές έχουν αποστείλει τις εκκλήσεις τους για διορισμού της ε, επιτροπές και Αντιπροσωπίας. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις στα πρακτικά της σημερινής ημέρας θα εγκριθούν αυτές οι προτάσεις τους. Οι αρμόδιες αρχές της